Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να καλωσορίζω 150 μαθητές και μαθήτριες από 33 ε, χώρες. Καλωσορίσατε στη Γιουροσκόλα είναι μια διημερίδα από χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και την Ουκρανία στα πλαίσια της Euroscola Euronest και θα συζητήσουν θέματα που ε, ενδιαφέρουν την ανατολική γειτονία. Είναι καλό να βλέπει κανείς νέους να συμμετέχουν στο δημοκρατικό γίγνεσθε. Και είναι μακρύς ε, ο ο διάλογος από τη δημοκρατία μέχρι την ε, εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συζητήσεις που είχατε. Ήταν πάρα πολύ ζωντανές, ε, με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος συμμετείχατε εκεί και ε, δεν υπολείπεται σε τίποτα η δική σας συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σε εύχομαι καλή επιτυχία στη ζωή σας και τη σταδιοδρομία σας επαναλαμβάνεται η σύνοδος, η περίοδος σύνοδου που ε, διακόπη στις 24 του μηνός Οκτωβρίου. Ο Σάνφος Τίερ έχει μια ερώτηση, παρακαλώ. 100.000 iz vukovarske bolnice do memorijalnog groblja najvee masovne grobnice u europi. Ε, έκαναν πορεία στο Βούκοβα ε, και ε, είναι 22 χρόνια μετά τη μάχη. Για πρώτη φορά, από τότε που είναι μέλος η Κροατία, έρχεται αυτή η επέτειο της μάχης του Βούκοβα. Γι' αυτό ήρθε και ένας αριθμός Κροατών πολιτών σήμερα στο ημικύκλιο επισκέπτες και θα ήθελα εξ ονόματός σας να τους χαιρετήσουμε, να τους καλωσορίσουμε και να αποτίσουμε το σεβασμό μας στους πεσόντες στη μάχη του Βούκοβα. Τώρα έχει έρθει η ώρα να ζούμε όλοι σε μια ενωμένη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στία για τα όσα μας είπατε και την υπόδειξη αυτή. Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 24 Οκτωβρίου διατίθενται. Έχετε στάσεις, αντιρρήσεις, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα συνοπτικά πρακτικά. Ερχόμαστε στις ανακοινώσεις. Οι αρμόδιες αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας με ενημέρωσαν για την εκλογή της κυρίας Γκαμπριέλη στα